και του δημοσίου χρέου των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλοι συνάδελφοι ανεφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να ασχοληθεί με αυτό, προκειμένου να μπορέσουν όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στη σημαντικότατη αυτή πρόκληση χρηματοδοτικά. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είναι υψηλέ οι φιλοδοξίε μα όσον αφορά την οικολογία και το περιβάλλον, όσον αφορά την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, θα πρέπει να βοηθήσουμε όμω όλε τι περιφέρειε, ακόμα και τι πιο ευάλωτε. Θα πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε περισσότερο στην αντιμετώπιση του κλίματο για να καταφέρουμε να φέρουμε το μέρο μα στου Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Χόρντι Κάνια για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπη, στη διάρκεια της κρίσης ένας φίλος οικονομολόγος ε, μου έλεγε ότι πίσω από τα μακροοικονομικά μέτρα που εγκρίνονται υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι. Του έλεγα εγώ μάλλον και μου λέει ας πάμε πιο πέρα. Ε, η βιωσιμότητα όπως ε, και ε, οι κρίσεις είναι κάτι που το πληρώνουν οι πιο ευάλωτοι και ο δρόμος, το μονοπάτι προς αυτό, η μετάβαση δεν θα πρέπει να την πληρώσουν και αυτή τη φορά οι πλέον αδύναμοι και ευάλωτοι. Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια Ευρώπη πιο βιώσιμη αλλά και πιο δίκαιη και υπάρχουν ορισμένοι που βάζουν μπροστά από το βιωσιμότητα κάποιε έννοιε και ιδέε που ξεχνάνε ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπου που είναι από πίσω. Χρειάζονται κονδύλια, ναι, πράγματι, αλλά χρειάζονται και στόχοι και αξίε. Οι αξίες αυτές ε, θα πρέπει να καθοδηγούν ε, τι πολιτικέ μα και πρόκειται για την κοινωνική πολιτική, για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα. Και μιλάμε για συγκεκριμένου στόχου. Ε, για να αγγιθούμε στου συμπολίτε μα ότι ποτέ πια δεν θα έχουμε κρίση, μετάβαση, αλλαγή που θα την πληρώνουν οι πλέον ευπαθεί, οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτε μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ερνέστ Ουρτασούν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Συζητούμε το επενδυτικό πρόγραμμα, το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, που θεωρώ ότι είναι σημαντικά στοιχεία του Νεοπράσινου Συμφώνου. Για το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, ε, τα είπαν και οι σύντροφοι, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά θα οδηγήσει σε μια μετάβαση. Άρα η αιρεσιμότητα να φύγουμε από τον άνθρακα και να ε, καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή είναι ένα στόχο και πρέπει να ενταχθεί αυτό το στοιχείο. Είναι κεντρικό στοιχείο στο Ταμείο Δίκαιη Μετάβασης για να μην μείνει κανεί πίσω πίσω. Είναι λοιπόν καλό που έχουμε αυτή την προτεραιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο των βιώσιμων επενδύσεων, από ό,τι ξέρουμε, νιώθω ότι δεν έχουμε επαρκή φιλοδοξία για να έχουμε και επαρκή πόρου. Αυτό το ε, σχέδιο Juncker 3.0, ε, κάτι τέτοιο μου μυρίζεται και μάλιστα κατεψυγμένο. Επομένω, ε, πρέπει να βρούμε νέε πηγέ χρηματοδότηση για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Λυπάμαι που αμφιβάλλω αν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το ποσό. Και γι' αυτό σα παρακαλώ παρακαλώ να είστε πλέον φιλόδοξοι για να είναι αυτό το σχέδιο πραγματικά ένα εργαλείο για μετασχηματισμό. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παόλο Μπόρκια για, για ένα λεπτό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα επηρεαστούν περίπου 500.000 εργαζόμενοι. Πάρα πολλοί είναι οι πόροι που χρειάζονται επίσης για το νέο αυτό πρόγραμμα, το οποίο προωθείται σαν νέο Ευαγγέλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια στρατηγική Απομάκρυνση από τη χρησιμοποίηση άνθρακα που όμω οδηγήσει μόνο στην αύξηση τη ανεργία και σε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλούμεθα όλοι να ακολουθήσουμε εντελώ μυρολατρικά το δρόμο αυτό που μα χαράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν δρόμο από βιομηχανοποίηση. Το περίφημο αυτό Ταμείο Δίκαιη μετάβαση. Χίλια δισεκατομμύρια ακούσαμε, μα δεν υφίστανται τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Είναι εντελώ θεωρητική η πόρη αυτή. Πιστεύω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να συγκεντρώσουμε τους του πόρου αυτού, θα καταφέρουμε πραγματικά να μετεκπαιδεύσουμε όλου αυτού του εργαζόμενου που θα χάσουν τη θέση εργασία του. Θα ήθελα πραγματικά να με εξηγήσετε πώ θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό στην πράξη. Πώ θα εφαρμοστεί σε μια χώρα σαν τη δικιά μου, την Ιταλία, που δεν υπάρχουν καν τα χρήματα αυτά. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Αναζελεύσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ακόμη και υπέρμαχοι ε, της πρότασής σας λένε ναι μεν αλλά. Και λένε αλλά γιατί το προτινόμενο σχέδιο είναι πολύ επιφανειακό. Δεν αρκεί να λέμε θέλουμε και υποσχόμαστε. Ε, θα, βέβαια το 2014 οι χώρες ε, συμφώνησαν για να μειώσουν τις εκπομπές κατά 30%. Και όλοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέχρι στιγμής που πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Ε, έχω ερώτηση, γιατί είναι πολύ επιπόλαια αυτά τα νούμερα που μας υποβάλλεται και που ε, προκαλούν την ε, απλή μαθηματική λογική. Είπατε ένα τρισεκατομμύριο, από πού θα βρεθούν όλα αυτά και πώς θα φτάσουμε στα 100 δις που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ένα που έχουμε τώρα. Με νέες επενδύσει, θέλω πιο συγκεκριμένε πληροφορίες, πιο λεπτομεριακέ. Επίσης, ε, θέλετε 300 δις από τους ε, ιδιώτες επενδυτές. Πώς όμως θα τους προσελκύσετε. Πότε επίσης θα έχουμε το νέο κλιματικό σύνταγμα. Ε, γιατί μόνο 60 μέρες έχουμε. Μας έχουν απομείνει. Ο κύριος Πέτερ Λίζη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα την Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ε, καλό αυτό το όραμα ε, της κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη και ήδη το 2018 ε, είχε δείξει το δρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αύξηση των θέσεων εργασίας και με την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται και κάποιες συνθήκες, κάποιες προϋποθέσεις, ένα πλαίσιο. Και είναι καλό που έχουμε αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης γιατί θέλουμε όλοι να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι και αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις περιφέρειες. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε για το νέο στόχο παλαιά κριτήρια και ε, στις πλούσιες περιφέρειες υπάρχουν ε, πολλές ε, απαιτήσεις για τον κόσμο που ζει εκεί και έχει να κάνει με την απαλλαγή από τον άνθρακα. Χρειάζεται σίγουρα εθνική υποστήριξη, αλλά θα πρέπει να εγκρίνει τα μέτρα αυτά στήριξης και η Κομισιόν. Με το ETS επίσης θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη αντίσταση επαρκής για τα όσα προτείνονται σε ό,τι αφορά το ETS. Τώρα, ε, ένας συνάδελφος ε, που κάθεται πίσω μου ε, λέει κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σωστά. Δεν θα είχαμε, κύριε Τίμερμαν, αν δεν ήσασταν εδώ, αυτήν την, το Ταμείο. Και ελπίζω να το πετύχουμε και στρέφομαι και στους συναδέλφους από εδώ που έχουν βοηθήσει. Ο κύριος Ντανίκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρότασή σας για τα 7,5 δις που θα πρικοδοτήσουν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Επίσης, χαιρετίζω και την πρωινή ανακοίνωση, δηλαδή το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει σχέδια που θα οδηγήσουν την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απαλλαγή της από τις εκπομπές άνθρακα. Ε, στη Ρουμανία είναι απαραίτητο όλα αυτά. χρειάζονται πάνω από 80 δις που θα χρειαστούν. Πάνω από 4% του ΑΕΠ θα είναι οι αιτήσεις δαπάνε που χρειαζόμαστε για τη δίκαιη μετάβαση και χωρίς την υποστήριξη της ΕΤΕΠ θα είναι αδύνατο να ανταποκριθούμε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι στιγμής στήριξε και βοήθησε τις πιο εύπορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνέβη στο παρελθόν και ελάχιστα βοήθησε τις χώρες που έκριζαν μεγαλύτερη ενίσχυση. Θα ήθελα να επιμείνω λοιπόν τα πιο απαραίτητα προγράμματα για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα να ξεκινήσουν αμέσως. Επίσης χρειάζονται κοινωνικά προγράμματα σε αυτές τις περιοχές και περιφέρειες, γιατί στην Ρουμανία, για παράδειγμα, πολλοί κάτοικοι θα επηρεαστούν από τέτοια σχέδια. Ο κύριος για ένα λεπτό. Καλημέρα σας. Προέρχομαι από μια χώρα, τη Γαλλία, όπου οι πολίτες φορούσαν ε, εδώ και πάρα πολλέ εβδομάδε κίτρινα γυλαίκα για να τονίσουν ότι ακριβώ η οικολογική μετάβαση θα πρέπει να είναι μια δίκαιη μετάβαση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η πρώτη πολιτική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής μετά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το Ταμείο και ο μηχανισμό δίκαιη μετάβαση. προκειμένου καμία ευρωπαϊκή επικράτεια να μην μείνει στο περιθώριο, προκειμένου κίνδυνοι να γίνουν ευκαιρία. Απευθυνόμενο στου συναδέλφου από την άκρα δεξιά που διαδέχονται ένα στον άλλον για να πούνε ότι θα μα κοστίσει πάρα πολύ, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό και το καθεξής. Μα πείτε πραγματικά, πηγαίνετε να δείτε του πολίτε από την Βενετία και ρωτήστε του πραγματικά αν θεωρούν ότι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την κλιματική αλλαγή. Απευθύνεται επίση το ίδιο ερώτημα στου πολίτε τη Αυστραλία. Πείτε του, θεωρείτε ότι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή ή μήπω το ότι δεν έχουμε αναλάβει επαρκή δράση αυτή τη στιγμή οδηγεί σε μια καταστροφή του ίδιου του πλανήτη μα. Αυτή είναι η πραγματικότητα πραγματικότητα. Ας ατενίσουμε λοιπόν το μέλλον και στο κάνουμε αυτό από κοινού και είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Μην ανησυχείτε, έχετε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δέχεστε μία ερώτηση, ρωτάει η Πρόεδρο, στο πλαίσιο τη διαδικασίας τη Γαλάζιας καρτα Η κυρία Βυσνιεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, Είστε ευρωβουλευτή από τη Γαλλία. Και πραγματικά με ευνηδιάσατε με τα σχόλιά σας. Εδώ και μήνε στη Γαλλία διαδηλώνουν τα κίτρινα γυλαίκα κατά τη κλιματική πολιτική. Το ενεργειακό σα μείγμα μόνο κατά 2% ε, στηρίζεται στον άνθρακα, ενώ το ε, πολωνικό ενεργειακό μείγμα 80% εξαρτάται από τον άνθρακα τι τεράστιο κόστος θα έχει μια τόσο περιοριστική κλιματική πολιτική για το πολωνικό έθνος. Μια δίκαιη κλιματική και ενεργειακή μετάβαση δεν θα πρέπει να αγνοεί τη φωνή του λαού. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση και εμεί το υποστηρίζουμε και εγώ προσωπικά το υποστηρίζω, ακριβώ επειδή σε χώρε όπω η δική σα, η Πολωνία, το σημείο κίνηση, το σημείο αφετηρία είναι διαφορετικό. Και χαιρετίζω αυτή τη στιγμή το γεγονό ότι η Πολωνία δεν μπλοκάρισε την, τον στόχο τη κλιματική ουδετερότητα. Θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό η κυβέρνησή σα και δεν το έκανε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή ελληνική, προκειμένου να έχουμε και στην Πολωνία μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Παντού στην Ευρώπη και ιδίω σε εσά. Σε καμία περίπτωση λοιπόν εγώ δεν είπα το αντίθετο. Υποστηρίζω το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση ακριβώ επειδή δεν αφήνει στο περιθώριο καμία χώρα και καμία περιφέρεια, ιδίω στι περιοχέ εκείνε και τι χώρε εκείνε που το έχουν ιδιαίτερα ανάγκη όπω η Πολωνία. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ράσμους Άντρεσεν. Για ένα λεπτό. πρέπει να δώσουμε απαντώσεις ε, ε, για τους ε, ακτιβιστές των 20 ετών, για τους 50χρονους ανθρακορίξου από την Πολωνία, για πολλά θύματα επίσης καρκίνου. Και σίγουρα θέλουμε μια δική μετάβαση για τις περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα μέτρα για την ανακύκλωση. Θέλουμε 25% επενδύσεις ε, για το κλίμα. Ε, να κάνουμε περισσότερα ε, σε σχέση με όσα ξεκίνησαν ο κύριος Γιόνκερ και ο κύριος Έτιγκερ, διότι δεν μπορούμε μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε το πράσινο σύμφωνο. Δεν θα φροντίσουν οι, οι ΕΡΒΕ και άλλοι όμιλοι ενεργειακοί, διότι τα θύματα θα είναι πρώτα αυτοί οι 50χρονοι ανθρακορίχοι και οι υπόλοιποι. Ε, θέλουμε επίσης Google, Amazon να πληρώνουν τους φόρους τους και να συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ε, και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση και των, διοξι... εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από άλλες χώρες. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό πιδελταπή και θα είμαστε και επιτυχείς. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ιζαμπέλα Ελένα Κλότς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Για πολλές χώρες μέλη ε, το, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο είναι οι μοναδικές πηγές ενέργειας στον δρόμο για την ε, κλιματική ουδετερότητα. Η Συμφωνία των Παρισίων ε, στηρίζεται στην ανάγκη χρήσης ιδίων πόρων για την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης τη, της ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να εκμεταλλευτούμε και τον άνθρακα και τα ανθρακοριχεία μας. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω από όλα τεχνολογική ελαστικότητα και χρόνο για να υλοποιήσουμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Για μας ε, ε, μόνο από το 2070 και μετά θα καταφέρουμε την κλιματική ουδετερότητα. Και τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι εμπειρογνώμονε θεωρούν ότι μια άκαμπτη περιβαλλοντική πολιτική θα οδηγήσει σε δυνητικό blackout στην Ευρώπη το 2050. Επίσης, ε, θα υπάρξουν σημαντικές ε, απειλές στην υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχουν ε, αρκετά, σχόλια, αρκετά πορίσματα που να αποδεικνύουν την επικινδυνότητα του άνθρακα, γιατί μπορούμε να έχουμε και πιο φιλικές προς το προβάλλον χρήσης του άνθρακα. Ε, εδώ, ε, χάρη στον άνθρακα, τον πολωνικό άνθρακα, σώζεται η ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας σε πολλά πράγματα. Θέλουμε λοιπόν ένα δίκαιο ταμείο μετάβασης ε, και κυρίως να είμαστε ειλικρινεί απέναντι στους συμπολίτε μας. Η κυρία Γκράσα Καρβάλιο, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά υιοθέτησε μια φιλόδοξη θέση για την κλιματική μετάβαση και την περιβαλλοντική προστασία. Για να υλοποιήσουμε όμως αυτή τη φιλοδοξία θα πρέπει από την αρχή να εξασφαλίσουμε δύο στοιχεία. Καταρχήν, οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις κλιματικές και περιβαλλοντικές μας προτεραιότητες και δεύτερον, οι επενδύσεις μας θα πρέπει να είναι αντάξιες των φιλοδοξιών μας και να μην γίνουν εις βάρος των ε, τρεχουσών πολιτικών και των ε, διαφόρων δημοσιονομικών γραμμών. Ε, επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και διασυνοριακής μετάδοσης γνώσης. Χρειαζόμαστε ένα απλό και ευέλικτο σύστημα κρατικών ενισχύσεων για να πραγματοποιήσουμε τη δίκαιη μετάβαση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες και ειδικέ ανάγκες κάθε περιφέρειας και επίση να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη τι περιφέρειε που θα έχουν τι μεγαλύτερε δυσκολίε στη μετάβαση. Κανέναν οικονομικό κλάδο δεν θα πρέπει να αφήσουμε ουραγό. Επίση, να μην ξεχνούμε ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκονται άνθρωποι. Ο άνθρωπο θα πρέπει να βρίσκεται ανέκαθα στο επίκεντρο τη στρατηγική μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριο Χώνα Φερνάντε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω τους αντιπροέδρους της Κομισιόν, να ευχαριστήσω και τον κύριο Τίμερμανς που αναφέρθηκε στην Αστούρια, στη δική μου την περιφέρεια, στη Βόρεια Ισπανία που εδώ και δεκαετίες ε, πλήττεται από το 1980 αρχικά όταν είχε να αντιμετωπίσει την απαραίτητη προσαρμογή μετά την πετρελαϊκή κρίση δεκαετία στα 70 και που σήμερα πλήττεται εκ νέου αντιμετωπίζουμε μια νέα πρόκληση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Στη δική μου την περιφέρεια αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουμε αντιληφθεί την αναγκαιότητα να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή αλλά ως σοσιαλιστές θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει βαθμιδών, να είναι ισορροπημένη και να εγγυάται ε, ισότη μεταχείριση όλων των συμπολιτών. Γι' αυτό ζητώ, ε, μάλλον θέλω πω ότι είναι καλή αυτή η πρόταση ως βάση διπραγμάτευσης για την εκκίνηση των συζητήσεων. Σίγουρα μένουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που θα πρέπει ακόμη στην διαδικασία τη νομοθετική να προσδιοριστούν Πρέπει επίσης ε, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ε, ε, συντομότερα, ένα φόρο προσαρμογή στα σύνορα των άνθρωπων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέρνερ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την πρόταση για ένα πράσινο σύμφωνο και ένα ταμείο μετάβασης και νομίζω ότι επιτέλους πια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σθένος και αισιοδοξία την ανάγκη την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής με καινοτομία, με φάνταστο τρόπο και όχι με ε, σχεδιασμένη, προγραμματισμένη οικονομία και με απαγορεύσεις ε, ή επιβολή καθηκόντων και υποχρεώσεων. Και για όλα αυτά πρέπει επίσης να προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως αυτό προβλέπεται. Δεν θα το καταφέρουμε με το ε, ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο χωρίς την συμμετοχή ιδιωτών ε, ως επενδοτών. Σίγουρα πιστεύω ότι η ΕΤΕΠ μπορεί να βοηθήσει και αυτό θα φροντίσουμε να κάνουμε και από πλευρά Γερμανία. Ό,τι αφορά τον συνάλφο Ράιλ που μίλησε για την κοιλάδα του Ρουρ και την σχετική περιοχή, δυστυχώ δεν είναι εδώ, αλλά ω ε, βουλευτή από την Βόρεια Βεσφαλία πρέπει να πω ότι η κατάσταση είναι τελείω διαφορετική σε αυτή την περιοχή. Γιατί εδώ και δεκαετίε δεν μπόρεσε να υπάρξει ε, η απαραίτητη αναδιάρθρωση και μόνο με συνεχείς ενισχύσεις. Το θέμα είναι πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο για ένα νέο μέλλον, να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να αλλάξει δουλειά. Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε τα μάτια μας στην κλιματική αλλαγή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Πέτρα Ντεσούτερ. Για ένα λεπτό. Και σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σαφώς η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί σημαντικότατη πρόκληση. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λάβει χώ, να αντιμετωπιστεί γρήγορα και θα πρέπει βέβαια να γίνει με τρόπο δίκαιο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακοίνωσή της. Θα πρέπει να βρεθούν όμως και απαραίτητη χρηματοδότηση. Η δίκαιη μετάβαση έχει ως στόχο να βοηθήσει τις περιοχές εκείνες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται πάρα πολύ από τα ρηκτά καύσιμα. Δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν όμως οι περιφέρειες εκείνες οι οποίες απλώς δεν θέλησαν όλα αυτά τα χρόνια να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα μολονότι θα μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτείτε μια δύσκολη συμφωνία με απρόθυμα ορισμένε φορές κράτη-μέλη. Μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια, έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Και πιο σημαντικά, αν κατακλείδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση να γίνει υπό προποθέσει. Τα κράτη-μέλη που θα λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν και συγκεκριμένε επιδόσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένα σχέδια απομάκρυνση από τον άνθρακα για καταπολέμηση κλιματική αλλαγή. Η κυρία Γιατιβίκα Βυσνιεύσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σήμερα ακούσαμε το νεφελώδες και πολύ γενικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με το Ταμείο Δικαιής μετάβαση και το προτινόμενο ποσό σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί γιατί ε, μόνο κατ' όνομα μάλλον θα είναι ε, δίκαιης μετάβαση στο Ταμείο. Και μάλιστα ρωτήσαμε τι θα γίνει με τις ε, ανθρακοπαραγωγές ε, ε, περιοχές της Πολωνίας. Και είπε ο αρμόδιος επίτροπος ότι ξέρει θα πονέσει αυτό το θέμα στους ανθρακορίχους. Οπότε πώς θα υλοποιήσουμε εμείς τη δίκαιη μετάβαση δεν θα πρέπει ε, το κόστος της, δημο... της ε, μετάβασης να το πληρώσουν μόνο οι ανθρακοπαραγωγές περιοχές και οι ανθρακορύχοι. Όπως η πατρίδα μου, η Πολωνία, που έχει πολλές περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Πριν ο συνάδελφος εγκομίασε το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών, αλλά... Πού βρίσκεται η δίκη μετάβαση αφού έχουμε τόσο διαφορετικές ενεργειακές τιμές. Ποιο είναι το κόστος της ε, κλιματικής ιδιαιτερότητας, πόσο θα κοστίσει αυτό στην Πολωνία που το ενεργειακό της μείγμα κατά 80% εξαρτάται από τον άνθρακα. Τι κονδύλια μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε χρόνο και χρήμα στην Πολωνία για να υλοποιήσουμε την κλιματική ουδετερότητα. Η Ursula von είπε ότι η κλιματική πολιτική δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω. Ελπίζω να τηρήσετε την υπόσχεσή σας. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Το λόγο έχει η κυρία Ισαμπέλ Μπεχουμέα Μπεχουμέα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση για το πράσινο σύμφωνο. Συμφωνίε για την προστασία του περιβάλλοντο ε, δεν μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτε βλάβε ε, στην οικονομία και πολίτε. Υπάρχουν ε, κάποιε συμφωνίε για να πετύχουμε την απαλλαγή από τον άνθρακα. Και τώρα πρέπει να θετήσουμε μέτρα ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικά και να δημιουργούν ευκαιρίε για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Είναι λογικό λοιπόν οι ευρωπαϊκέ περιφέρειε που θα πληγούν την απαλλαγή από τον άνθρακα και, για την, και από την μετεγκατάσταση του κλάδου θα χρειαστούν αντιστοιχιστικά μέτρα. Η Ισπανία, ε, οι περιοχέ με τα θα πληγούν. Δεν είναι λογικό ένα κράτος μέλος ε, το οποίο τηρεί παρέγκλητα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να θυγεί επειδή έκανε αυτό που έπρεπε. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς και γιατί. Το Ταμείο Δίκης Μετάβασης πρέπει να βοηθήσει τις στιγμόμενες περιφέρειες ε, να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές, να ανακυκλωθούν, να μετατραπούν οι κλάδοι σε κάτι πιο προσοδοφόρο για το μέλλον. Δεν θα πρέπει ε, ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για να ε, έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας. Ε, επίσης θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του στόχου, του προορισμού, του αποτελέσματος των επενδύσεων, συγκεκριμένα σχέδια που θα ε, συνηγορούν υπέρ της ε, εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της αναζήτησης σε πιο, πιο ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Άγνες Γιονχέριους. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να υλοποιήσουμε πρόοδο και κοινωνική μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον οδικό χάρτη για την κοινωνική Ευρώπη. Βέβαια, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, αλλά η πρόθεση του χάρτη είναι ξεκάθαρη. Κανένα δεν θα πρέπει να μείνει ουραγός ή στο περιθώριο. Ξέρουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση θα φέρουν πολλές αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε νέες θέσει σε νέα ταμεία και χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να πραγματοποιήσουμε μια βιώσιμη μετάβαση και δίκαιη ταυτόχρονα. Ε, επίσης, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια κονδύλια της ε, ΚΑΠ και όπου και αν εργάζεται κάποιος, ακόμη και σε πλατφόρμα, να προσβλέπει σε έναν αξιοπρεπή, ε, αξιοπρεπή μισθό. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ένα δίκαιο μισθό, δίκαιε αμοιβέ και για του εργαζόμενου σε πλατφόρμες Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταπολεμήσει και την κλιματική ένδυα, γιατί θα είναι δύσκολη η υλοποίηση τη δίκαιη μετάβαση υπάρχει τέτοια διάσταση απόψεων στο Συμβούλιο, τόσο διαφορετικά σχέδια εθνικά, θα πρέπει να βρούμε κάποια χρήματα και για την κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Χαϊτάμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες. Οι πυρκαγιές, οι καταστροφικές στην Αυστραλία καταδεικνύουν με τον πλέον πρόδειλο τρόπο ότι θα πρέπει να λάβουμε δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Πράσινα Συμφωνία πρόκειται να λειτουργήσει μόνο αν την εστερνιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχει κανένα νόημα η συμφωνία αυτή αν φτάσουμε σε τέτοιο σημείο ενεργειακή ένδυα που οι Ευρωπαίοι πολίτε θα μπορούν καν να πληρώνουν του λογαριασμού του αν δεν μπορεί η ευρωπαϊκή καινοτομία να οδηγήσει σε τεχνικέ οι οποίε θα μα βοηθήσουν στο μετριασμό τη κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν η υποστήριξη και ο σχεδιασμό μα να είναι μακροπρόθεσμα και θα πρέπει να μπορέσουμε να αντλήσουμε πόρου και μέσω τη ευρωπαϊκή φορολογία. Αντί όμω να ζητήσουμε ευθύ αμέσω χρήματα από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, μήπω θα ήταν καλύτερο να έχουμε την πολιτική, αν θέλετε, αξιοπρέπεια και να δούμε τελικά πού μπορούμε να απελευθερώσουμε χρήματα από τον κοινοτικό προπολογισμό, δίνοντα ένα νέο προσανατολισμό σε κάποιε πολιτικέ προτεραιότητε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει καταρχά να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν την κοινοτική του χρηματοδότηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προτού ζητήσουν νέα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η, η κυρία Καρολίν για ένα λεπτό. Η εφαρμογή του Ταμείου της Δίκης Μετάβασης είναι ένα καλό μαντάτο γιατί μία μετάβαση θα είναι επιτυχής μόνο αν είναι ακριβοδίκαιη ε, κοινωνικά και ισο, ισο, ε, ίση. Ε, επίσης, ε, έχουμε το κλάδο του άνθρακα που εκπέμπει πολλές ε, ανθρακούχες εκπομπές. Επίσης, ε, οι μερυπογόνε δραστηριότητε βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομίας και είναι σημαντικός, πολλές φορές, σημαντική πηγή ε, απασχόλησης και εισοδημάτων. Δεν θα πρέπει να καταλήψουμε στη μοίρα τους αυτούς τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να τους δώσουμε βιώσιμες ευκαιρίες, να τους ε, ανακυκλώσουμε σε νέες ε, θέσει απασχόληση ε, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια ή στην κυκλική οικονομία. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την υποστήριξή μας στις περιοχές που θα κάνουν την μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσαρμοστούν στον τόχο ε, του Παρισίου, τη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης, θα πρέπει ε, να μην χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο για να, για να χρηματοδοτήσουμε άλλες ε, ενέργειες ορυκτές όπως το ε, αέριο και να έχουμε ένα είδος αιρεσιμότητας. Είναι σημαντικό να απεμπλέξουμε, να απελευθερώσουμε κονδύλια για την επιτυχία της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση για τα θέματα αυτά. Το λόγο ο κύριος Κρίστιαν Σίλβιο Μπουσόη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα μόνο μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης θα καταφέρουμε να ε, πετύχουμε όλα τους, όλους τους στόχους που έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης θα καταφέρουμε τελικά να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όντως να διασφαλίσουμε την υποστήριξη αυτή Ας μην ξεχνάμε ότι ένα 41% των περιφερειών της Ρουμανίας θα επηρεαστούν από την ε, πολιτική κλιματικής αλλαγής της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφώ τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να περάσουμε στην νέα αυτή φάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και για να καταφέρουμε να προωθήσουμε μια οικονομία πιο ψηφιακή. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βρούμε φρέσκο χρήμα και να μην παίρνουμε χρήματα από το Ταμείο Συνοχή. Η κυρία Κωνσταντσε Κρέλιχ, τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επικροτώ την πρόταση της Κομισιόν για το Πράσινο Σύμφωνο και την πρόταση για το Ταμείο Δικής Ανάπτυξης, ε, Δίκης Μετάβασης. Είναι εξαιρετικές οι προτάσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο δύο σε αυτές τις περιφέρειες που θα θυγούν. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία, για τα οποία θα ήθελα κάτι περισσότερο. Πρώτον, το θέμα της χρηματοδότησης. 7,5 δις ε, για το ETF, ε, αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Ε, δεν θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να χρησιμοποιηθούν παλαιά κονδύλια. Νέο ναι, νοπό χρήμα θέλουμε. Δεν μπορούμε να περικόψουμε τα κονδύλια της συνοχής και δεν μπορούμε τελικά με αυτό το ταμείο ε, να στερήσουμε περιφέρειες από τη χρηματοδότησή τους και για το ε, ΔΕΛΤΑΠΗ ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση. Η πρόταση του Συμβουλίου είναι χειρότερη, κατώτερη από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Πρέπει να προετοιμάσουμε την μετάβαση, όχι να στηρίζουμε ανέργους όμως, αλλά να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για άτομα που έχουν ακόμη δουλειά. Ευχαριστώ. Το λόγο για ο κύριος ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και τα κονδύλια για το Ταμείο Δίκης Ανάπτυξης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αλλά οφείλουμε να το πραγματοποιήσουμε. Γιατί στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το πρόγραμμα Invest in Europe. Υπολογίζεται ότι η πολιτική συνοχής απορροφά ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού. Ένα τμήμα της χρηματοδότησης θα πρέπει να διοχετευτεί και στη δική μετάβαση και να χρηματοδοτήσουμε κυρίως τις περιφέρειες εκείνες που ήταν πολύ εξαρτημένε από τον άνθρακα και το κλείσιμο των ανθρακοριχείων του θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη, την, τον εξυγχρονισμό βιομηχανικών τεχνολογιών για να εγκαταληφθεί σταδιακά ο άνθρακα. Έτσι θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας με χαμηλή χρήση άνθρακα. Κύριος Μπλος. Για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόφσκι, κύριε Τίμερμαν, πραγματική προστασία του κλίματο δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη γι' αυτό και είναι πολύ θετικό που έχετε λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή και όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε και να επενδύσουμε σε νέε θέσει εργασία για το μέλλον, για πιο φιλοπεριβαλλοντικέ θέσει εργασία. Αυτά τα οποία έχετε καταθέσει όμως ως προτάσεις μέχρι τώρα είναι πολύ λίγα. Δεν ε, προτείνεται νοπό χρήμα, αλλά ουσιαστικά αλλαγή ε, και μεταπίδηση κάποιων κονδυλίων σε άλλους ε, τομείς. Πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από τον άνθρακα. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει και με την υποστήριξη από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Γερμανία θέλει προστασία του κλίματος χωρίς να θέσει ε, γι' αυτό παραπάνω κονδύλια. Δεν πρόκειται αυτό να λειτουργήσει. Ε, δεν έχουμε ποτέ πετύχει κάτι με μηδενικά κονδύλια ή μόνο με ωραία λόγια και υποσχέσεις σε ε, ευχολόγια. Χρειαζόμαστε κλίμα, ε, πρακτική προστασία, αλλά και δικαιοσύνη κλιματική και πρέπει να είμαστε συνεπεί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Άνταμ Γιαρούμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Α, νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πρωτοφανείς α, προκλήσεις ε, και υποσχέσεις παγκοσμίω ε, για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και μάλιστα είχαμε κάποιε αλλαγέ σε σχέση με του στόχου του 2030. Οι αλλαγέ που προτείνουμε θα απαιτήσουν το μετασχηματισμό ολόκληρη τη οικονομία και όχι μόνο τον ενεργειακό ανασχηματισμό. Και αυτό θα έχει τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Γι' αυτό θα πρέπει η μεταμόρφωση αυτή, αυτός ο μετασχηματισμός να είναι δίκαιος, η μετάβαση να είναι δίκαιη και με ικανοποίηση διαπιστώνουμε το στόχο του Ταμείου Δικής Μετάβασης και την δημιουργία του. Φυσικά το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει κατεξοχήν τις ε, ε, περιοχές που θα έχουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, για την μετάβαση, την ενεργειακή μετάβασή τους και θα έχουν και τις πιο δαπανηρές διαδικασίες τέτοιας μετάβασης με μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ που θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτό. Επίσης, ε, ε, το κονδύλιο που προτείνεται ελπίζουμε να είναι η αρχή και στο μέλλον να πρικοδοτηθεί και με νέα κονδύλια το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ίσως και με ίδιους πόρους ε, όπως ο φόρος του άνθρακα ή άλλοι φόροι της κοινής αγοράς. Ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Μαργαρίτα Μάρκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ταυτόχρονα υπέβαλε αυτά τα τρία έγγραφα στα πλαίσια της γενικής της στρατηγικής. Οι κλιματικές αλλαγές δημιουργούν ανισότητες και οικονομικές και κοινωνικές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το αναγνωρίσει και να δράσει για να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει αυτές τις ανισότητες. Περιμένουμε λοιπόν αντίστοιχε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Βέβαια, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και αερίου του θερμοκηπίου. Οπότε θα είναι δυσανάλογη η μετάβαση των κρατών μελών. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει ψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γιατί έδωσε προτεραιότητα στη φιλοδοξία των ΑΠΕ και έχει επενδύσει ε, σημαντικά ποσά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να, να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε όλες τις περιοχές ε, χωρίς εξαίρεση για την ενεργειακή τους μετάβαση, να προωθούμε τον εξυγχρονισμό της οικονομίας τους και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Πορ Χόλμγκρεν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώ η πρωτοβουλία αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντική, με σαφώ υπέρ επίση μια δίκαιη μετάβαση. Τάσουμε λοιπόν υπέρ των προτάσεων αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να λάβουμε δράση και όχι γενικά και αόριστα στο μέλλον. Αναφερόμαστε όμω πιο συγκεκριμένα σε ένα ταμείο δίκαιη μετάβαση, μία από τι τρει προτάσει που μα έκανε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες εκείνες οι οποίες θα λάβουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρούν βέβαια και τους στόχους τους κλιματικούς, έτσι δεν είναι αν είναι να χρηματοδοτήσουμε χώρες οι οποίες έχουν οικονομίες που βασίζονται στον άνθρακα, τότε θα πρέπει πραγματικά οι χώρες αυτές να αρχίσουν να προσανατολίζονται σιγά σιγά προς άλλες πηγές ενέργειας και να απομακρύνουν όλο και περισσότερο από τον άνθρακα. Θα πρέπει οι χώρες αυτές να δημιουργήσουν πράσινε θέσει απασχόληση και να έχουν νέε μορφέ οικολογική πράσινη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να θέσουμε του Ευρωπαίου πολίτε στο κέντρο τη κλιματική μα πολιτική. Μόνο τότε η προσπάθειά μα θα στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ κύριο Μπούζεκ. Ένα λεπτό. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μου για την υποβολή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συγκεκριμένες προτάσεις στήριξης των περιοχών που περισσότερο ε, τη χρειάζονται αυτή την υποστήριξη. Έχουμε επιτάπητος πολλές προτάσεις, μπορούμε να τις συζητήσουμε. Και πιστεύω ότι χάρη στις προτάσεις θα έχουμε μια θετική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των προτάσεων και έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε όλες τις συναφείς εκθέσεις. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θεσπίζεται ώστε οι πολίτες, κυρίως στις πλέον απειλούμενες περιοχές, να πιστούν ότι η κλιματική ουδετερότητα το 2050 θα υλοποιηθεί μαζί με τους πολίτες, χάρη των πολιτών και όχι εις βάρος των πολιτών. Και ιδιαίτερα στις ανθρακοπαραγωγές περιοχές. Για παράδειγμα, ε, στο Κατοβίτσε έγινε η COP24. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη υποστήριξη αυτή η περιοχή που εξαρτάται από τον άνθρακα. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια και τη χρηματοδότηση του Ταμείου μετάβαση. Μετάβασης. Θα πρέπει να βρούμε συμπληρωματικά κονδύλια. Γι' αυτό σκεφτείτε το κύριε Αντιπρόεδρε. Πού θα βρούμε επιπρόσθετα κονδύλια, όχι μεταφορά κονδύλιων από άλλε πολιτικές. Θέλουμε νοπό χρήμα ε, και νέα κονδύλια που θα βρουμε επιπροσθετα κονδυλια οχι μεταφορα κονδυλιων απο αλλε πολιτικε θελουμε νοπο χρημα και νεα κονδυλια που θα πρεπει να γράψουμε στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μουνίρ Σατουρί για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και για το χάρτη πορεία για την κοινωνική Ευρώπη, λυπάμαι που δεν έχουμε εδώ πέρα τον Επίτροπο Σμίτ. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφαιρθούμε και στην προστασία των δημοσίων υπηρεσιών στην ε, προστασία των θέσεων απασχόλησης, στην προστασία των ανθρώπων ε, των άστεγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά αποτελούν πτυχές της δίκαιης μετάβαση και μιας κοινωνικής Ευρώπης. Παντού στην Ευρώπη έχουμε σημαντικότερες ανισότητες οι οποίες επιδεινώνονται. Η υπερθέρμανση του πλανήτη επίσης ε, επιτείνει τι σημαντικότερε αυτέ ανισότητες οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται από την άκρα δεξιά για να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη μα. Χρειαζόμαστε περισσότερε δεσμεύσει όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Και επαναλαμβάνω εδώ πέρα ότι εμεί οι οικολόγοι περιμένουμε ακόμα περισσότερε δεσμεύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η οικοδόμηση αυτού του κοινωνικού πυλώνα να γίνει μια πραγματικότητα για όλου του Ευρωπαίου πολίτε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Φραντ Μπογκόβιτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρώπη αποφάσισε να ανταποκριθεί στην, ε, ευρωπαϊκή, στην κλιματική έκτακτη ανάγκη. Έχουμε λοιπόν ως απάντηση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που έρχεται όμως με ένα τίμημα. Ενώπιό μας λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία πρόταση για έναν μηχανισμό και ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης. Σαφώς είμαστε υπέρ των πρωτοβουλειών αυτών. Θα πρέπει να προασπίσουμε τις πιο ευάλωτες περιοχές, όπως για παράδειγμα τον τομέα των ανθρακοριχών στην ε, Πολωνία. Σαφώ θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές, αλλά δεν είναι οι μόνες οι οποίες θα καταβάλουν ένα σημαντικό το τίμημα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επομένω, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι προκειμένου να καλύψουμε και όλες αυτές τις νέες υποδομές που θα απαιτηθούν για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές, για να καταφέρουμε να αποζημιώσουμε και άλλους τομείς οικονομίας, όπως για παράδειγμα το τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι τομείς πολιτικής που θα πρέπει να καλυφθούν από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει στα πλαίσια του πλαισίου αυτού να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα στοιχήσει το Ταμείο Αυτοδίκαιης Μετάβασης και πού θα βρεθούν τα χρήματα. Ο κύριος Ατμαρκάρας. σε ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε θέσει σωστούς δικαιούς στόχους, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αρκετά φιλόδοξη η στόχη αυτή. Επίσης γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο μονομένο μέτρο που θα μπορέσει να εφάρμοσει από μόνο του τους στόχους αυτούς. Χρειάζονται πολλά λιθαρά και χρειάζονται διάφορες προσεγγίσεις ε, και χρειάζονται και χρήματα. Και γι' αυτό είναι και σημαντικό να έχουμε 260 εκατομμύρια το χρόνο ως επενδύσεις και χαιρετώ ε, αυτό το ποσό που προτείνεται ε, ε, ενός τρεις για την επόμενη δεκαετία. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και να καταφέρουμε να πετύχουμε πρόοδο. Και καλό είναι να έχουμε και αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, διότι υπάρχουν κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές που θα πληγούν περισσότερο και πρέπει να να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα, ε, για να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και να σταθεροποιήσουμε τις περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό το κοινωνικό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε, αλλά υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να τις αναφέρουμε και να τις αναγνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέρμπερτ Τόρφμαν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως ε, χρειάζεται ενεργειακή μετάβαση, ότι χρειαζόμαστε πρώτες ε, ε, και λιγότεροι σε εκπομπές του του άνθρακα και πολλοί από τους συναδέλφους ε, είπαν πολύ σωστά ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να καθορίσει και καθορίζει τα ανθρακοριχεία που κλείνουν, ε, τις αλλαγές επίσης του πολιτική και εκεί έγκυται και η απώλεια θέσεων εργασίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εργαστεί ε, στα ανθρακοριχεία και χρειάζονται νέες ε, προοπτικές, αλλιώς δεν ε, θα έχουν μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε προς το μέλλον, να βρούμε προσεγγίσεις, παραδείγματος να ενισχύσουμε τη βιοτεχνολογία, να βρούμε εναλλακτικέ πρώτε και έχουμε και αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που δεν πρέπει απλά να είναι ένα ταμείο το οποίο θα φροντίσει ε, να αποζημιωθούν όσων τα δουλειέ χαθούν, αλλά είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να δημιουργεί και νέε προοπτικέ και νέε θέσει. Ευχαριστώ. Το λόγο και ο κύριο Λεβαντόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και μόνο το όνομα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ε, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική κατανομή και δίκαιη κατανομή των κονδυλίων. Δίκαιη δηλαδή ανάλογα με το βάρος που φέρει κάθε περιοχή με το άχθος της ε, ενεργειακής μετάβασης. Και αυτό ισχύει περισσότερο για τις ε, ανθρακοπαραγωγές περιοχές που για ιστορικούς λόγους ε, ήταν ανέκαθεν εξαρτημένες από τον άνθρακα. Γι' αυτό και η Νέα Πράσινη Συμφωνία μας βρίσκει σύμφωνος. Ναι, μεν, αλλά, γιατί η Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι μόνο πράσινη, αλλά και ανταγωνιστική. Ναι, μεν, αλλά για να η ηγηθεί του κόσμου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει επιτυχή πολιτική περιβαλλοντική και να μην είναι παταγώδης αποτυχία. Και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε ε, τις αδρές γραμμές αυτής της πολιτικής. Προς το παρόν είναι ομιχλώδης η κατάσταση. Ε, μόνο όταν δούμε συγκεκριμένες προτάσεις θα μπορούμε όλοι με μία φωνή να πούμε «Ναι, μπορούμε, yes, we can». Νομίζω ότι κύριε και κύριοι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν ακόμη 35 ε, προτάσεις, ετήματα για τη διαδικασία προσέγγισης προσοχής του Προέδρου και ε, γι' αυτό δεν μπορώ λόγω και των συζητήσεων που έπονται να δώσω το λόγο παρά μόνο σε 8 συναδέλφους ε, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Επόμενη είναι η κυρία Μαρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσετε το μηχανισμό για τις βιώσιμες επενδύσεις και τη δίκαιη μετάβαση έχει ιδιαίτερη σημασία να λάβουμε υπόψη ότι για να πετύχει ο μηχανισμός για τη δίκαιη μετάβαση οφείλουμε να καθορίσουμε άμεσα τα κριτήρια επιλεξιμότητας με γνώμονα τη συνεισφορά της παραγωγής του άνθρακα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής αλλά και την ταχύτητα της απομάκρυνσης από τον άνθρακα στην ελλάδα η κυβέρνηση μέσω του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα έχει ήδη ανακοινώσει ότι επιχειρεί να κλείσει τις μονάδες του άνθρακα έως το 2023 και πάντως το ενεργειακό μείγμα της ελλάδος δεν θα προέρχεται από τον άνθρακα το. 2028. ή όχι η ταχύτητα της απανθρακοποίησης ένα στοιχείο για την επιλεξιμότητα στο ταμείο δίκαιης μετάβασης; αντιπρόεδρε τίμερμανς σας άκουσα να αναφέρεστε στους πολίτες της δυτικής μακεδονίας. περιμένουν εδώ από εμάς στο στρασβούργο και τις βρυξέλλες να τους δώσουμε μια δίκαιη προοπτική να αντικαταστήσουμε την αγωνία τους με μια βιώσιμη δουλειά δουλειές που τους ταιριάζουν δουλειές για τη βιομηχανία δουλειές για τη ενέργεια. περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Εντίνα Τότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Είμαι υπέρ τη απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Αυτό θα απαιτήσει όμω πόρου, χρηματοδότηση και περαιτέρω επενδύσει. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν παρουσιάζουν ακόμα σημαντική οικονομική ανάπτυξη, που έχουν τι χαμηλότερε αποδοχέ και αυτέ που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα και εκεί όπου θα χαθούν θέσει απασχόληση. Μέσω του Ταμείου Δίκαιη Μετάβαση μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το ενεργειακό κόστο ή το κόστο τροφίμων δεν θα αυξηθεί στι περιοχέ αυτέ. Σαφώ δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε καμία περιοχή και θα πρέπει η μετάβαση αυτή ενεργειακή να είναι δίκαιη και ισότιμη. Το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση, λοιπόν, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τι παραδοσιακέ δημοσιονομικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να πάρουμε χρήματα από τι ήδη φυστάμενε πολιτικέ. Χρειαζόμαστε νοπό χρήμα, νέου πόρου εκτό του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Α μην ξεχνάμε ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο για τι χώρε αυτέ που θα πρέπει να απαλλαχθούν από τον άνθρακα. Κύριο Σόκολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, οι, αλλαγές είναι πραγματικό... οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το βλέπουμε και παγκοσμίω και στην Ευρώπη. Στην πατρίδα μου την Κροατία, για παράδειγμα, ε, οι παράκτιες πόλεις ε, το Ζάνταρ, το Σπλί, το Ντούμπροβνικ είναι πραγματικά κοσμήματα πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Θα πρέπει να δούμε όμως και τις συνέπειες της ενεργειακής μετάβασης, τις κοινωνικές και τις οικονομικές. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξή. Όταν μιλούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη συμφωνία, ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε μια σημαντική αξιολόγηση των συνεπειών των προτάσεων. Επίσης, ε, να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι χρήσεις μεγαλύτερης προστασίας περιοχές. Τρίτον, θα δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή μετάβαση και να μην γίνει η χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, που είναι η σημαντικότερη πολιτική αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική συνοχή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περικοπούν τα κονδύλια της. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι κονδύλια θα χρηματοδοτηθεί η δίκαιη μετάβαση και με τι κριτήρια θα γίνει η κατανομή των κονδύλιων. Μέχρι στιγμή, δυστυχώς όλα αυτά δεν διευκρινίζονται. Ευχαριστώ. Λίντια Περέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι στόχοι της νέας πράσινης συμφωνίας είναι μια πιο αναπτυγμένη, πιο εχής Ευρώπη με βιοπικιλότητα, ε, και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με μια κυκλική οικονομία που θα προωθεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. η Είναι αναμφίβολο ότι η μετάβαση αυτή είναι και περιβαλλοντική αναγκαιότητα αλλά και οικονομική ευκαιρία. Το σχέδιο βιώσιμη επένδυση είναι ένα σχέδιο που δίνει σάρκα και οστά στι φιλοδοξίε μα και λέει ότι 25% του κοινοτικού προπολογισμού θα διορθωθεί στο στόχο τη ε, ενεργειακή μετάβαση δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, βιώσιμες επενδύσεις και επενδύσεις σε νέες ιδέες και τεχνολογίες. Αυτά είναι τμήματα στρατηγικής που θα φέρει την Ευρώπη ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο ως ηγέτη με μια ανταγωνιστική και ανεπτυγμένη οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στις ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως την ηλιακή ενέργεια, αλλά και στη χρήση του υδρογόνου. Ε, έτσι θα λύσουμε άπαξ και διαπαντός τα προβλήματα ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης και των ισιωτικών περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Ο Σον Κέλλη δεν είναι εδώ. Ο κύριος Κούλογλου. Λόγος εδώ και μήνες για το μηχανισμό δίκαιας μετάβασης και τις προσδοκίες που υπάρχουν γι' αυτό Σήμερα ακούσαμε στοιχεία και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Εγώ θα ήθελα να σα υπενθυμίσω πω στην Ελλάδα οι περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι θα πληγούν από το κλείσιμο των μονάδων στην περιφέρεια Δυτική Ελλάδο και το Δήμο Μεγαλόπολη. Στην Ελλάδα δεν ακούμαστε σε ένα απλό recovery από την απερχόμενη, όπω όλα δείχνουν, κρίση, αλλά στοχεύουμε σε μια μεγάλη ελληνική πράσινη έκπληξη. Δεν αρκεί να λέμε σε ένα οργανισμό, σε μια περιφέρεια να πρασινίσει πρέπει να τις δείχνουμε τον τρόπο και να τις παρέχουμε τα εργαλεία χωρίς να αποδυναμώνουμε επιτυχείς δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει στην πραγματικότητα ο μηχανισμός να είναι όχι μόνο δίκαιης, αλλά και αποτελεσματικής μετάβασης. Θα πρέπει να αποδείξουμε στους ανθρώπους που θα αλλάξουν αντικείμενο εργασίας ότι δεν θα χάσουν τι δουλειέ του και ότι υπάρχει ένα όχι μόνο εθνικό ή τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό σχέδιο που θα διαφυλάξει τι επενδύσει, τι επιχειρήσει και το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε περιοχή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κίμπουρόπλο ήταν και όχι ο κύριο Κούλογλου. Ο κύριο Ρουίθ Ντεβέσα. Ε, Λόπες Λόπεθ Κύριος Αγγιλάρ. Κυρία Βόρντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στην απομακρυσμένη μου περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που γενιές ανδρών και αγοριών σαν δούλοι δούλευαν κάτω στα ανθρακοριχεία ε, για να δημιουργηθούν εξαρτήματα για πλοία, για σιδηρόδρομους και πολλά χιλιάδες άλλα προϊόντα. Βοήθησαν λοιπόν τις υποδομές, βοήθησαν τη βιομηχανία και το εμπόριο και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται όταν εξαφανίζεται έτσι με μια κίνηση αυτή αυτή βιομηχανία. Στη μεταβιομηχανική Αγγλία και μετά την κυβέρνηση της Θάτσερ στον Τάραμ οι ανθρακορίχοι το μόνο που κατάφεραν να έχουν είναι χαμηλά αμοιβόμενες δουλειές στις γραμμές παραγωγής 7 μέρε ε, τη βδομάδα ασχολούνταν με το να βάζουν παραδείγματο χάρη πατατάκια στι σακούλε. Ε, και πραγματικά ήταν άνθρωποι που έχασαν την αξιοπρέπειά του. Ε, και τι διαφορά θα είχε γίνει αν υπήρχε τότε για αυτούς τους άνδρες, για αυτά τα αγόρια της περιφέρειάς μου, το Ταμείο Δίκης Μετάβασης. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι. Ξέρουμε ότι έχουμε υπέρβαση ωραρίου. Είχαμε 35 αιτήματα και ε, από τους ε, πέντε που έχω εκφωνήσει ένας είναι παρόν ε, μέχρι τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ, μόνο χρόνο δαπανούμε όταν εγώ πρέπει να ρωτάω κάθε φορά ποιος είναι και ποιος δεν είναι παρόν από όσους έχουν ζητώσει. Μπάρμπαρα Γκίψον είναι η επόμενη στον κατάλογο. Δεν είναι εδώ. Σουσάνα Σόλες Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση. Το Ταμείο Δικής Μετάβασης έχει θεμελιώδη σημασία για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και για να χρηματοδοτήσουν την απαθρακοποίησή τους. Μιλούμε για ένα τρισεκατομμύριο ευρώ σε μία δεκαετία. Θα δούμε όμω πώ θα κατανεμηθούν τα διάφορα κονδύλια. Κύριε Τίμερμαν, εσεί στην παρουσίασή σα αναφερθήκατε στου ανθρακορίκου τη Αστούρια, τη γενετηρά μου. Αλλά και η Καστιγελαιών, η Αστούρια, η Αραγωνία είναι περιοχέ που έκλεισαν τα ανθρακοριχεία του, έκαναν το καθήκον του και τώρα κλείνουν και τα τελευταία εργοστάσια παραγωγή άνθρακα που εξαρτώνται ε, Παραγωγή ηλεκτρισμού συγγνώμη, που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Αυτό όμω έχει πειράσει πολύ την απασχόληση και οδηγήσει στην απερίμωση των περιοχών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω να λάβετε υπόψη αυτέ τι περιοχέ που έκαναν το καθήκον του, να μην τι ξεχάσετε στο Ταμείο Διοικητική μετάβαση. γιατί όπω είπατε δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν ουραγό ε, και είναι σημαντικό να μην χαθούν και άλλε θέσει απασχόληση ε, και του κατοίκου του οι περιοχέ αυτέ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκταν Ρόντσα. Ευχαριστώ. Ζόντσα, συγγνώμη. Ε, στα θέματα της ταξινόμησης ε, α, αναφέρθηκε, κανονισμό ένα παραθυράκι για το φυσικό αέριο που αναφέρεται ως μεταβατικό, μεταβατική ενεργειακή πηγή. Αναφέρεται έτσι τουλάχιστον στην πρόταση. Κύριε Επίτροπε, ε, πώς εννοείτε εσείς την μεταβατικότητα ε, του φυσικού αερίου. Ε, γιατί ε, είπε άλλος επίτροπος ότι δεν θα περικοπούν οι τρέχουσες επενδύσεις, δεν θα διακοπούν οι τρέχουσες επενδύσεις, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο. Και ξέρω ότι δεν είναι κλιματικά ουδέτερο, αλλά σίγουρα είναι ένα ασφαλές μέσο ενέργειας, μια ασφαλής πηγή ενέργεια. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πιο θετικοί απέναντι στο φυσικό αέριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μάρκ Ποτέγκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση που μας έγινε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία επί τα οποία θα ήθελα να σταθώ. Αν πραγματικά θέλουμε μια δίκαιη μετάβαση, τότε θα πρέπει να εστιαστούμε και στο ζήτημα των δημοσίων υπηρεσιών θα υποστηρίξετε, μα είπατε, τι τοπικέ αρχέ. Για ποιο λόγο όμω να μην καταργήσετε μια και καλή τη πολιτική λιτότητα, Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουν οι απαραίτητε δημόσιε επενδύσει για να μην κλείσουν, για παράδειγμα, οι μικροί σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.ο.κ. Το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να θέσετε επίση στι διαπραγματεύσει που κάνετε είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού τάμπινγκ. Εσεί λέτε ότι θα πρέπει απλώ να εφαρμοστούν οι φυστάμενοι κοινοτικοί κανόνε. Μα θεωρείτε ότι υπαρκεί αυτό, ε, όχι προφανώ. Και τρίτον, όσον αφορά την απασχόληση, μα είπατε ότι θα υποστηρίξετε κυρίω τι μεγάλε επιχειρήσει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μα το πρόβλημα είναι ότι αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Του δίνουμε επιδοτήσει, του δίνουμε ενισχύσει, περιμένουμε από αυτέ να κάνουν κάτι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Τα λοιπόν τα χρήματα αυτά και προχωρούν. Ο κύριος Πάτεν έχει το λόγο. Απουσιάζει. Μάντερς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση αποτελεί μια σημαντικότητα πρόκληση, γιατί βλέπουμε ότι όλοι θέλουν χρήματα και όλο και περισσότερα χρήματα. Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον πάντω η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα γίνει ένα εξαγώγημο, αν θέλετε, προϊόν. Κάτι το οποίο θα μπορέσει να προωθήσει προς τα έξω